ήσυχα από την αίθουσα. Να ξεκινήσουμε με τις επεξηγήσεις ψήφου. Έκθεση HEAD. Πρώτο στον κατάλογο η κυρία Όβερ. Φαίνεται ότι έχουμε πρόβλημα με το μικρόφωνο της κυρίας Οβίρ. Παρακαλώ, μιλήστε τώρα. Ε, ja, Νύτ on ε, Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την προστασία των καταναλωτών τη σχετική πολιτική της και τη ρυθμιστική της πολιτική έχει αλλάξει πολύ τις κινήσει και τι ενεργές τη τα τελευταία χρόνια. Έχει ε, προαχθεί ιδιαίτερα και το ηλεκτρονικό εμπόριο το τελευταίο διάστημα και βλέπουμε και τη σημασία των διασυνοριακών καταναλωτικών ε, συναλλαγών. Η προστασία λοιπόν των καταναλωτών γίνεται όλο και περισσότερο σημαντική, καθότι οι πολίτες ε, αγοράζουν και πολλούν ε, πέραν των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό να δείξουμε μεγαλύτερη ευελιξία στην πολιτική προστασία των καταναλωτών και στα ε, μέσα της και στηρίζω τόσο την έκθεση όσο και τις τροπολογίες όπως εγκρίθηκαν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπαλσίτης επόμενος. Thank you, ε, Mr. Chairman, colleagues. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, υπερψήφισα την έκθεση αυτή, διότι η ενίσχυση τη πολιτική προστασία των καταναλωτών είναι καθοριστική σημασία για την λειτουργία, την λειτουργία τη εσωτερική αγορά. Θέλουμε μια τέτοια αγορά που να λειτουργεί επαρκώ και αποδοτικά και για του καταναλωτέ. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει απόλυτα σήμερα και υπάρχει ισχύουσα νομοθεσία, η οποία όμω δεν έχει ενισχυθεί καταλήλω από τα κράτη-μέλη με εθνικά μέτρα. Οι καταναλωτέ δεν αισθάνονται πάντοτε ασφαλεί, διότι δεν γνωρίζουν πάντοτε του κανόνε και σε πολλέ περιπτώσεις οι μηχανισμοί αντιστάθμισης δεν λειτουργούν αποδοτικά. Η Επιτροπή λοιπόν θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της ώστε τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν σωστά τις οδηγίες και οι πολίτες να είναι πλήρως πληροφορημένοι για τα δικαιώματά τους και να μπορούν να ασκήσουν και τα δικαιώματά τους στην πράξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα ερχόμαστε στην διεύθυνση Μπουρζόη. Ο πρώτος στο κατάλογό μου είναι ο κύριος Σπάτσκιτς. I'm sorry. Your microphone doesn't... Το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Ε, thank you, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Σεγητά, οι συνάδελφοι ε, στήριξα την και υπερψήφισα αυτήν την πολύ καλή πρωτοβουλία, ιδίω ως προς την ιδέα να ενισχυθεί το δίκτυο Solvit και οι εθνικές δράσεις. Θα πρέπει όμως να εξεύρουμε και την απαραίτητη χρηματοδότηση για να βεβαιωθούμε ότι τα εθνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι πύλες του ίντερνετ ε, στο διαδίκτυο καθώς και τα τηλεοπτικά δίκτυα θα προβάλλουν σωστά την ε, δράση και τη λειτουργία του δικτύου Solvit. Μπορώ να σας πω ότι ήδη εφαρμόζονται διπλά μέτρα και σταθμά και πολύ συχνά τα νομοθετήματα προβλέπουν διαφορετικές κυρώσεις για τις ίδιες παραβιάσεις. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, παρακαλώ, όσοι εξέρχεστε τις αιθούσεις, ε, κάντε ησυχία. Ο κύριος Αντωνιώτση. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Υπεψήφισα την έκθεση Μπουσόη, διότι θεωρώ ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Solving είναι θεμολιώδους σημασίας για να υπάρχει μια σαφής και διάφανη σχέση μεταξύ θεσμικών οργάνων, πολιτών και επιχειρήσεων, που είναι ένα από τα σεμελιώδη στοιχεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Solvit ε, αποδείχθηκε ένα πολύ χρήσιμο μέσο για να επιληθούν τα προβλήματα των πολιτών και των επιχειρήσεων που θέλουν να εκμεταλλευτούν πλήρους τις δυνατότητες που προσφέρει η αγορά. Πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχουν ακόμα φραγμούς στην εσωτερική τους νομοθεσία και αυτοί οι φραγμοί πρέπει να αρθούν. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε την επιπλέον χρωματοδότηση, την, το επιπλέον εξειδικευμένο προσωπικό και την αύξηση της ε, προβολής αυτής της υπηρεσίας, ακόμα και σε τοπικό επίπεδο, όπου θα μπορούσε να ε, αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας παρακαλώ, μπορείτε να κάνετε τις συζητήσεις σας εκτός αιθούσης, ώστε να μπορούν να γίνουν οι επεξηγήσεις ψήφου. Ευχαριστώ πολύ. The next is Mrs. Reutova, please. Η κυρία Ρόιτοβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ως ε, σκιώδης εισηγήτρια θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την ψήφο του, Με τη συντριπτική πλειοψηφία εγκρίθηκε η έκθεση για το Solvit. Έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα υποχρεωθεί να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη τη δική μας σύσταση. Οι πολίτες και οι επιχειρηματίες ωστόσο θα πρέπει να είναι πολύ καλά προφορημένοι και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, την άλλη ε, ε, ε, χρονιά του χρόνου δηλαδή να μας φέρει μια ε, πολύ καλή πρόταση, μια πολύ καλή έκθεση για τα πορίσματα και τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής. Ευχαριστώ. Mr. Yao. Okay. Ο κύριος Yao. Oh, sorry. Oh. I'm, I'm awfully sorry. Α, ζητώ συγγνώμη, Πρόεδρος, εγώ φταίω. Προχωρούμε τώρα στην έκθεση De Bruyne και ο ε, πρώτος ομιλητής εδώ είναι ο κύριος Καλινόσκι. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να εξηγήσω την ψήφο μου για την έκθεση της κυρίας Δεμπρούν. Θα ήθελα να την ευχαριστήσω για την έκθεσή της. Μας ανησυχεί όχι μόνο η ευημερία των ζώων, αλλά και των ανθρώπων. Θα θέλαμε να μειωθεί ο χρόνος αναμονής και μας ανησυχεί και η εξάπλωση της λύσας. Θα θέλαμε να υπάρχει ελεύθερη μετακίνηση, να λαμβάνουμε υπόψη και τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Ευχαριστώ και τώρα η κυρία Ρόιτοβα για την έκθεση Τεμπρούν. Κυρία Ρόιτοβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπερψήφισα για τη διάταξη για την παράταση της μεταβατικής περίοδου, για τις εξαιρέσεις για τα κράτη, διότι τα κράτη είπαν ότι δεν θα ζητήσουν περαιτέρω παράταση. Εδώ θα ήθελα να καθησυχαστούν οι σουηδικές, βρετανικές ε, ανησυχίες για τα ζώα συντροφιάς που μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα ε, εκτός των διαφορών κρατών. Εδώ υπάρχει κίνδυνος λύσας και άλλων ε, ασθενειών. Και πρέπει δυστυχώς να σκεφτούμε την κατάργηση των περίοδων αυτών παράτησης στο μέλλον. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταλαβαίνω το ενδιαφέρον των διαφόρων κρατών μελών που ε, πιέζουν ε, για παράταση της μεταβατικής περίοδου. Θα πρέπει όμως να προσέξουμε ε, το κόστος και ωφέλεια να έχουν κάποια αναλογία μεταξύ τους. Και νομίζω αυτή ε, τη στιγμή στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ανεπαρκέ. Γι' αυτό και απήχα κατά τη διάρκεια της ψηφοφορία. Αυτό που χρειαζόμαστε κυρίως είναι εξωτερική προστασία όταν πρόκειται για εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη ε, όλο και περισσότερη εναρμόνιση στο εσωτερικό της Ένωσης και για την προστασία των καταναλωτών που τελικά χάνει ε, τις αναφορές, τα σημεία αναφοράς όταν ισχύουν άλλα σε μια χώρα εισόδου και άλλα σε μια άλλη χώρα. Ευχαριστώ, κυρία Σινκλέρ. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι κατά της πρότασης, γιατί έρχομαι από το Ηνωμένο Βασίλειο και πιστεύω ότι ήδη έχουμε επαρκεί νόμου να αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα, ιδίω με το κίνδυνο τη λύσα που αυτή τη στιγμή πλήττει την Ιρλανδία. Δεν καταλαβαίνω γιατί επαναφέρεται μόνο σε γάτε, σκύλου και παπαγάλου η πρόταση αυτή. Και νηφίτσε. Ε, πριν από 25 χρόνια αναγκαστήκαμε να σκεφτούμε και να ξαναδούμε έκτοτε αυτούς τους κανόνες. Έκτοτε όμως πολλοί εκλογείς από το Ηνωμένο, Βασίλειο πιστεύουν ότι η διατάξη που εδώ προβλέπουμε και νόμοι δεν θα είναι λογική. Ε, ε, γεια σας κύριε Πρόεδρε. Ε, χαίρομαι που σας ξαναβλέπω κυρία Πρόεδρε. Ακούμε πολλά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ανακατεύεται με πολλά η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει λιγότερα και καλύτερα. Και τώρα ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Ποια ζώα μπορούν να κυκλοφορούν πού. Ε, η αναλογικότητα πού είναι. Υπάρχουν χώρες που είναι νησιά, που δεν έχουν χερσαία σύνορα και μπορούν κάλλιστα να βρουν λογικές ε, διμερείς ή και πολυμερείς συμφωνίες μεταξύ τους. Είναι ανάγκη οπωσδήποτε να ανακατευτούμε εμείς. Είναι καλύτερο να δημιουργήσουμε και άλλη επιπλέον γραφειοκρατία στα χέρια των ίδιων ε, ευφυών ανθρώπων που μας έχουν φέρει όλες τις κοινέ πολιτικές, τον προϋπολογισμό, ε, τη γεωργική πολιτική και όλο αυτό το κοινοτικό κεκτημένο. Μα αυτό ακριβώς το θέμα μπορούν να το χειριστούν τα κράτη-μέλη. Πάμε τώρα στην έκθεση Κοέγιο, η κυρία Οβίρ πρώτη. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο και πάλι ο στόχος της ζώνης Σέγγεν είναι η ελεύθερη μετακίνηση. Είναι παράλογο οι κάτοχοι θεωρήσεων μακράς διαμονής να έχουν περιορισμούς ε, στην ελεύθερη μετακίνησή τους στην περιοχή Σέγγεν. Τα άτομα με ε, θεωρήσεις μικρής διάρκειας μπορούν να μετακινηθούν πολύ πιο εύκολα. Υποτίθεται ότι σε ένα μήνα θα ε, ξεκινήσει ο κώδικας για τις θεωρήσεις. Ωστόσο, η ερμηνεία που δίνεται στα κράτη-μέλη είναι διαφορετική ως προς τον τρόπο των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό που μας ανησυχεί κυρίως είναι πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι καθημερινά και καθυστερήσεις που διαπιστώνονται στα κράτη-μέλη. Το θέμα είναι κατεπήγον. Ο κώδικας των θεωρήσεων, όπως σας είπα, θα τεθεί σε ισχύ πολύ σύντομα και ήθελα τέλος να πω ότι υποστηρίζω την ε, έκθεση. Η κυρία Ρόιτοβα. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ υποστήριξα την έκθεση αυτή ε, για τις ε, θεωρήσεις μακράς διαρκείας. Γιατί είπαμε, οι ερευνητέ, οι φοιτητέ και οι υπόλοιποι θα πρέπει να έχουν την ελευθερία των κινήσεών του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα όμω να ζητήσω την αλληλεγγύη σα προ την Τσεχική Δημοκρατία που ε, αγωνίζεται ε, μάταια απέναντι στη βούληση του Καναδά και στην άρνηση του Καναδά να προσαρμοστεί και να συμμορφωθεί με το σύστημα θεωρήσεων. Το ίδιο ισχύει και με την Ουγγαρία. Ο Καναδάς υποσχέθηκε ότι θα αλλάξει την νομοθεσία του. Ε, ζητώ συγγνώμη που καταχράστηκα τις προσοχή σας για να μιλήσω για αυτό το θέμα. Η κυρία Γκάλ. Τα όσα ακούσαμε στη διάρκεια της συζήτησης είναι για να διευκολύνουν τους κατόχους θεώρησης ε, μακράς διαρκείας από τρίτες χώρες για να μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. δημιουργείται πρόβλημα επειδή δεν εκδίδονται εγκαίρως άδειες ε, παραμονής ή κάποια κράτη-μέλη δεν εφαρμόζουν σωστά το ε, ευρωπαϊκό δίκαιο. Η Ουγγαρία απήχε της διαδικασίας διότι θεωρούμε ότι εφαρμόζουμε το σύστημα τη διαδικασια διοτι θεωρουμε οτι καταλήλως και είμαστε ιδιαίτερως αποτελεσματικοί στην έκδοση αυτών των αδειών παραμονής, αλλά θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερω προσεκτικοί με τους κατοίκους τρίτων χωρών που συνορεύουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να διαμένουν σε μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά θα πρέπει να υπάρχει και νομοθεσία σε ευρωπαϊκό και κρατικό επίπεδο που θα διευκολύνει την κατάσταση. Και τώρα για την ε, έκθεση Σοφή κυρία Υπάρχουν πολλά καλά στοιχεία σε αυτή την έκθεση, αλλά δεν μπορώ να υποστηρίξω την εισαγωγή ενός ε, κοινού ε, παγιωμένου ε, το, δασμού. Επειδή οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να επιλέξουν να συμμετέχουν ή να απέχουν του συστήματος, αυτή τη στιγμή δημιουργούνται προβλήματα. Το προτινόμενο CCCTB σημαίνει ότι θα κατανέμονται τα έσοδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, μια χώρα σαν τη δική μου, την Ιρλανδία, η οποία εξάγει πολλά προϊόντα, θα τιμωρείται διότι τα κέρδη θα προσμετρώνται βάσει των εξαγωγών και επομένω δεν θα έχουμε ελεύθερη μετακίνηση αγαθών. Αν χρησιμοποιήσουμε το CCCTB, ουσιαστικά τιμωρούμε τι χώρε εξαγωγού. Και κάτι τέτοιο θα ε, μειώσει τη δυνατότητα της Ευρώπης να προσελκύσει ξένες επενδύσεις, διότι μέσω κάποιου περίπλοκου τύπου ο οποίος μπορεί μόνο να υπολογιστεί αναδρομικά δεν θα μπορεί να υπολογιστεί καταλήλως ε, ε, το ποσοστό και δεν θα μπορέσουμε φυσικά να προσελκύσουμε ξένους επενδυτές. Και τέλος για την έκθεση του Χόμσταϊν πρώτος ο κύριος Καλανόφσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη συνάδελφο για την έκθεσή της, η οποία είναι, δίνει πολύ καλά στοιχεία για την οικονομική ανάπτυξη. Στηρίζω λίγο πολύ σχεδόν όλα όσα είπε και την ε, εφαρμογή του ε, κοινοτικού δικαίου στην, ε, σε ολόκληρη την κοινότητα κοινότητα. Είναι σημαντικό να λάβουμε μέτρα τη στιγμή αυτή τη χρηματοπιστωτική ε, κρίση και να αξιοποιήσουμε πλήρω όσε δυνατότητε μα δίνει η αγορά. Θα πρέπει όμω και τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του κρατικού επίπεδου να συνεργαστούν μαζί μα. Χρειάζεται λοιπόν μια ε, αρμονική επικοινωνία μεταξύ των δημόσιων αρχών, προκειμένου να έχουμε απλοποίηση διαδικασιών και όλα αυτά είναι πολύ ευχάριστες ειδήσει, ε, συμπεριλαμβάνοντα την άμεση μεταφορά των ευρωπαϊκών οδηγών στα κράτη-μέλη. Περισσότερα να γίνουν στο επίπεδο τη επικοινωνία για τα δικαιώματα των πολιτών, τα δικαιώματα των επιχειρήσεων, να έχουμε περισσότερη διαφάνεια και περισσότερο ανταγωνισμό. Ο κύριος Οσμπάτσκιτ. Oh, Πρώτα ο κύριος όχι εσεί, Στη συνέχεια εσεί. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Υποστήριξα την καλή αυτή πρωτοβουλία και πιστεύω ότι ε, θα είναι πολύ ωφέλιμη για τους λαούς μας. Ωστόσο, αν δεν έχουμε πολύ ε, καλά ρυθμισμένη και λειτουργούσα εσωτερική αγορά με καλό έλεγχο και παρακολούθηση, δεν πρόκειται ε, να βοηθήσουμε ποτέ τους παράγοντες της αγοράς, ανεξάρτητα από το μέγεθος ε, της επιχείρησης ή της ε, υπηρεσίας που παρέχει ή χρησιμοποιεί. Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν σαφείς κυρώσεις και να επιβάλλονται σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται παραβίαση των κανόνων. Επίσης, θα πρέπει να βελτιώνεται η ε, διεθνής ε, διαδικασία ε, διευθέτηση των διαφορών ή ο διεθνής διακανονισμός. Γιατί διαπιστώνουμε αυτή τη στιγμή ότι 8 στις 10 περιπτώσεις χωλαίνουν και τα εθνικά δικαστήρια ή οι διάφοροι μηχανισμοί διακανονισμών ακολουθούν λάθος διαδικασία. Τώρα εσείς κυρία Οβίρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με συγχωρείτε που προσπάθησα να πάρω το μικρόφωνο πρώτη προηγουμένω για να έχουμε μια σταθερή και καινοτόμο αγορά και ένα εύρωστο και υγιές οικονομικό περιβάλλον πρέπει να εργάζεται και να λειτουργεί σωστά η εσωτερική αγορά. Θα πρέπει όμως όνο οι κανόνες και οι διακανονισμοί να εγκρίνονται εγκαίρως και να υλοποιούνται από τα κρατημέλη. Η έγκριση νομοθετικών μέτρων θα απλοποιηθεί και ο έλεγχο από το Κοινοβούλιο επίση θα διευκολυνθεί εάν και τα εθνικά κοινοβούλια μπλέκονται στην αρχή τη όλη διαδικασία και μάλιστα συμμετέχουν ενεργά. Ε, στήριξα πλήρω την έκθεση αυτή και συμφωνώ μαζί τη. Ευχαριστούμε και τέλο η κυρία Ρόιτοβα. Κυρία Ρόιτοβα. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως περιμέναμε και οι τρεις ερωτήσεις για την εσωτερική αγορά εγκρίθηκαν από την Ολομέλεια. Ωστόσο, στην τελευταία τούτη έκθεση, οι πράσινοι και οι σοσιαλιστές ήταν κατά των τακτικών ελέγχων λειτουργίας ε, της εσωτερικής αγοράς, γιατί είπαν ότι αυτό δήθεν είναι απειλή στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι προδιαγραφές αυτές έχουν ένα κόστος και οδηγούν και σε υψηλότερο βιωτικό επίπεδο. Ε, στην Ευρώπη. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο η συγκήτρια έχει πρόβλημα με αυτό. Εγώ υποστήριξα και τις τρεις εκθέσεις. Διακόπτεται η συνεδρίαση, λέει η πρόεδρος, ως τις 3 το απόγευμα.